Είμαστε έτοιμοι για τις ψηφοφορίες. Απλουστευμένη διαδικασία για την έκθεση Ρέουλ σχετικά με την ε, ένταξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην ε, υπηρεσία, στη Διεθνή Υπηρεσία ε, για τις ανανεώσιμες ενέργειες. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται τώρα. Ψηφίσατε όλοι. C'è una parte che dice sì e Κάποιοι λένε ναι, κάποιοι λένε όχι. Ε, δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη έτσι. Adesso credo che abbiate votato tutti. Τώρα νομίζω ψηφίσατε όλοι. Bene, dichiaro chiusa la votazione. Πέρας της ψηφοφορίας. Votanti in totale 470. Εψήφισαν 478 υπέρ 453 kata κατά 13 αποχές 12. Εγκρίνεται η έκθεση. Ha chiesto la parola l'onorevole Casini. Ζήτησε το λόγο ο κύριος Καζίνη, παρακαλώ. Δεν πρόλαβα. Αν είχα προλάβει όμως θα υπερψήφιζα. Μάλιστα. Ωραία. Να προσμετρηθεί άλλη μία ψήφος λοιπόν. Αυτή του συναδέλφου Καζίνη. Λοιπόν, πάλι απλουστευμένη διαδικασία για την έκθεση Ντεκάστρο κατάργηση κάποιων αποχαιωμένων κανόνων του Συμβουλίου στον τομέα της ε, κοινή ε, γεωργικής πολιτικής. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται τώρα. tutti? Ψηφίσατε όλοι. Καλώς πέρας της ψηφοφορίας. Εψήφισαν 543. Υπέρ 542. Κατά μία ψήφος. Αποχή. Μη. Δεν. Συντριπτική πλειοψηφία. Βουλγαρική όπως τη λέμε εμείς. Βουλγαρική. Αλλά όχι στη σημερινή Βουλγαρία που είναι απόλυτα δημοκρατική χώρα. Της παλαιάς. Ecco, Ψηφοφορία σύμφωνα με απλουστευμένη διαδικασία για την έκθεση Δεκάστρο για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων για τι εργαστηριακές αναλύσεις. Ονομαστική ψηφοφορία. Avete votato tutti? Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εψήφισαν 577 υπέρ 534 κατά 29 αποχές 14. Εγκρίνεται η έκθεση. Έκθεση Hübner Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται τώρα. Εψηφίσατε όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. Εψήφισαν 604 υπέρ 579 κατά 13 αποχές 12. Εγκρίνεται. Ο Σάφος Μάρτιν θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, θα ήθελα να πω ότι και εμένα δεν λειτουργήσε η δική μου συσκευή και εγώ ήθελα να ψηφίσω ναι, να υπερψηφίσω. Α, Σημειώνουμε. Κύριε Μαρτίν, τα λεγόμενά σας. Πάμε στο επόμενο πάντα προσθεμένη διαδικασία, Γκέριγκερ, για τα άγρια πουλιά. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Votanti 619, favorevoli 590. Ψήφισαν 619, υπέρ 592, κατά 4 αποχές 23. Εγκρίνεται η έκθεση Γκέρινγκ. Δεύτερη έκθεση Γκέρινγκ. Πάντα με απλωστευμένη διαδικασία. Ε, εξοπλισμοί που λειτουργούν με φυσικό αέριο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. 638, favorevoli 618. Ψήφισαν 638 υπέρ 618 κατά 11 αποχές 9. Εγκρίνεται η έκθεση Γκέριγκερ. Τρίτη έκθεση Γκέριγκερ για την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Άρχεται η ψηφοφορία. Avete votato tutti? La votazione è chiusa. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Εψήφισαν 641 υπέρ 620 κατά 13 αποχές 8 εγκρίνεται η έκθεση. Τέταρτη έκθεση Γκέριγκερ. Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας. Απλουστευμένη διαδικασία, άρχεται η ψηφοφορία. Avete votato Πέρα της ψηφοφορίας. Votanti 654 favorevoli 643. Ψήφισαν 654 υπέρ 643, αποχές 11, ψήφι κατά 0. Συγχαρητήρια κυρία Γκέριγκερ για, τρί, για τέταρτη φορά. Πέμπτη έκθεση Γκέριγκερ, πάντα πλουστευμένη διαδικασία. Κτηνιατρική έλεγχη των ζώων που προέρχονται από τρίτες χώρες. που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Εψήφισαν 657, υπέρ 644, σαν κατά 11, δύο αποχές. Εγκρίνεται. Έκτη έκθεση Γκέριγκερ. Δίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης επί των και της οικονομικής λειτουργίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων απλουστευμένη πάντα διαδικασία και ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινά τώρα που ολοκληρώνεται τώρα εψήφισαν 657 υπέρ 632 κατά 17 αποχές 8 εγκρίνεται 7η έκθεση Γκέριγκερ όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκινητές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επόαση. Από τρίτες χώρες ε, θέτω σε ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία την έκθεση. Κιούσα. Πέρασε ψηφοφορία. Ψήφισαν 662 υπέρ 641 κατά 15 Έξι αποχές. Εγκρίνεται και αυτή η έκθεση. Όγδοη έκθεση Γκέριγκερ σχετικά με τα καθαρόαιμα βοηδή αναπαραγωγής. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τις ψηφοφορίες. Ψήφισαν 655 υπέρ 633 κατά 13 9 αποχές. η συνάδελφος Γκέριγκερ έφερε σε αίσιο πέρας εννέα εκθέσεις, σχεδόν ρεκόρ. Παρακαλώ, χειροκροτήσατε. Περνάμε τώρα στον κύριο Μπουσουτήλ. Σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Μαυρικίου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχία διανομή. Αποσταμένη διαδικασία, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορίες. Ψήφισαν 662 υπέρ 602 κατά 32 28 αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερη έκθεση Μπουσούτιλ για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϊχελών για απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρηση για βραχία διαμονή. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες. Ψήφισαν 667, υπέρ 610, κατά 28, αποχές 29. Εγκρίνεται η έκθεση. Τρίτη έκθεση Μπουσουτήλ. Συμφωνία απαλλαγή για την υποχρέωση θεώρηση για βραχία διαμονή μεταξύ κοινότητα και Μπαρμπάντο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Ψήφισαν 663 υπέρ 604 κατά 29 αποχές 30. Εγκρίνεται και η τρίτη έκθεση Μπουσουτήλ. Πάμε στην τέταρτη έκθεση Μπουσουτήλ. Πάλι απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρηση για βραχία διαμονή μεταξύ κοινότητα και Αγίου Χριστόφορου και Νέβη. Άρχεται η ψηφοφορία. La votazione è chiusa. Votanti 660. Πέρα τη ψηφοφορία ψήφισαν 664 υπέρ 603 κατά 28, 33 αποχέ. Εγκρίνεται η έκθεση. Σουτήλ e approvata. Πέμπτη έκθεση Μπουσουτήλ. Συμφωνία για απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης μεταξύ κοινότητας και Αντίγουα και Μπαρμπούντα. Άρχεται η ψηφοφορία. <laughs> Μπαρμπούντα, ε, είπα, όχι Μπάρμπα, δηλαδή η γενιάδα του κυρίου Σούλτς, έτσι. Πέρα της ψηφοφορίας. Ψήφισαν 672, υπέρ 612, κατά 29, αποχές 31. Εγκρίνεται. Έκτη έκθεση Μπουσούτιλ σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχία διαμονή και την αντίστοιχη συμφωνία μεταξύ της κοινότητος και α, την Βρετανική Κοινοπολιτεία. Τις Μπαχάμες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Ψήφισαν 672 υπέρ 608 κατά 31 αποχές 33 εγκρίνεται και αυτή. Συγχαρητήρια κύριε Μπουσουτήλ. Για την έγκριση, για την υιοθέτηση έξι εκθέσεών σας στην συνεδρία αυτή της Ολομελίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πάμε τώρα στην έκθεση Χάουγκ διορθωτικός προπολογισμός υπαρθμών 9 του 2009 για τον σεισμό στην Ιταλία. Άρχεται η ψηφοφορία, χρειάζεται ειδική πλειοψηφία. Votazione è chiusa. Πέρα Votanti ψηφοφορία. Ψήφισαν 673 υπέρ 654 κατά 4 αποχές 15 εγκρίνεται η έκθεση Χάουγκ. Ευχαριστώ κυρία Χάουγκ και στο όνομα της Ιταλίας το λέγω αυτό. Πάμε τώρα στην έκθεση Μπόγκε για την κοινοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίησης. Ονομαστική ψηφοφορία χρειάζεται ειδική πλειοψηφία. Άρχεται η ψηφοφορία. La votazione chiusa. Πέρα τη ψηφοφορία. Ψήφισαν 677 υπέρ 598 κατά 49 30 αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Μπόγκα. Προβάτα. Πάμε στην έκθεση Wallis. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Μάρεκ Σίβιετσα. Άρχεται η ψηφοφορία. E chiusa la votazione. ψηφοφορία. Ψήφισαν 671 υπέρ 639 κατά 17, 15 εποχές. Εγκρίνεται η έκθεση. Έκθεση Κοέλιο. Μηχανισμός αξιολόγησης για την παρακολούθηση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σέγγεν. Δεν υπάρχουν τροπολογίες. Την θέτω λοιπόν την έκθεση ως έχει σε ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Stiamo votando la proposta di decisione sulla quale ψηφίζουμε για την πρόταση επί της οποίας δεν υπάρχουν τροπολογίες. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Όχι. Λοιπόν, καλά, εντάξει, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Ψηφίζουμε την πρόταση απόφασης yeah, επί είναι η γνωμοδότηση Κοέλιο και για την οποία δεν υπάρχουν τροπολογίες. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεν είναι ονομαστική. Δεν είναι ονομαστική η ψηφοφορία. Διανατάσσεω χειρό μπορείτε να ψηφίσετε. No, διανατάσεως χειρός ε, κύριε Σπερώνη. Παρακαλώ ψηφίσατε. Ε ποιος είναι υπέρ. Α, πρέπει να πω ποιος είναι υπέρ, ε. Ποιος είναι κατά. Έτσι <laughs> ε, voleva, voleva tanto, Allora, la relazione... Σαφές, σαφές απορρίπτεται η έκθεση. Μπορεί να Έχει τη δυνατότητα να ομιλήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλετε να διατηρήσετε την πρότασή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ναι, αν... να σηκωθείτε παρακαλώ. Ο συνάδελφός μου, ο κύριος Μπαρό, αντιπρόεδρος της Επιτροπής, τόνισε ότι οι προτάσεις αποβλέπουν στην κινητικοποίηση του μηχανισμού αξιολόγησης ούτως ώστε να γίνει ε, πιο αποτελεσματικός ενώ διατηρείται η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών. Η Επιτροπή είναι πεπισμένη ότι το Κοινοβούλιο ε, πρέπει ε, να συμμετέχει στην αξιολόγηση Schengen, πράγμα που δεν γίνεται τώρα. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων. Ωστόσο, βάσει των, των που ισχύουν δεν μπορούμε με συναπόφαση να εμπλέξουμε το Κοινοβούλιο ούτως ώστε να συμμετάσχει. Γι' αυτό διατηρούμε τις προτάσεις βάσει των, των γύρων συνθήκων. Όσο προς την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, ο φάκελος αυτός θα ξανανοίξει και η Επιτροπή θα αποφασίσει εν ευθέτω χρόνο ποια θεωρεί ότι είναι η κατάλληλη νομική βάση για το μηχανισμό που προτείνεται ούτως ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσει να συμμετάσχει όσο το δυνατόν περισσότερο. Η Κομισιόν ίσως ε, προτείνει ε, νέες προτάσεις τροποποιημένες ανάλογα με την περίπτωση. Καλώς. Ακούσατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να διατηρήσει την πρότασή της, άρα ε, παραπέμπεται απευθείας στην Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών. Παρακαλώ κύριε Κοέλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τις, ε, για τις διευκρινήσεις του τον κύριο Επίτροπο. Θα ήθελα όμω να επιθυμήσω, όπω κατέστησα σαφέ κατά τη διάρκεια τη συμφωνη... ότι η νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανεγνώρισε την νομιμότητα τη νομική βάση τη πρόταση τη Κομισιόν, αλλά είπε ότι από τη βάση τη ισχύωση συνθήκη είναι απόλυτα δυνατόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει λάβει την ίδια πρωτοβουλία επί τη βάση επί τη βάση άλλης νομικής, ε, άλλου άρθρου ως νομική βάση. Για μεγαλύτερη δηλαδή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό προτείνω η πρωτοβουλία να επανέλθει, το θέμα να επανέλθει σε εξέταση στην Επιτροπή και να μπορέσει να αναθεωρήσει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το χρονικό διάστημα προβλέπεται από το άρθρο 55 του καταστατικού μας μπορούμε να αναμένουμε μια νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που να σέβεται την συναπόφαση και που να δώσει σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την αναγνώριση που χρειάζεται για να μπορέσει να υπερασπίσει τα δικαιώματα του πολίτου στα πλαίσια του, χώρου, ε, του κεκτημένου του χώρου Σέγγεν. Ευχαριστώ κύριε Κοέλιο. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε από αυτού που είπατε, γιατί αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να διατηρήσει επιτάπητο την πρότασή τη. Η πρόταση αυτή αυτομάτω παραπέμπεται στην Επιτροπή, όπω ακριβώ ζήτησε ο συνάδελφο Κοέλιο. Περνάμε στην δεύτερη έκθεση Κοέλιο για την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που θεσπίζει ένα μηχανισμό αξιολόγησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου Σέγγεν. Πρόκειται για πρόταση κανονισμού επί της οποίας δεν υπάρχουν τροπολογίες. Την θέτω σε ψηφοφορία. Δεν χρειάζεται ονομαστική ψηφοφορία. Υπέρ παρακαλώ. Ποιος είναι κατά, ποιος απέχει, τέλος πάντων δεν χρειαζόταν αυτό το τελευταίο γιατί είναι σαφές ότι απορρίπτεται η πρόταση. Έχει τον λόγο ο Επίτροπος. Ναι κύριε Επίτροπε, είναι ίδια περίπτωση και συνεπώς η θέση της Επιτροπής είναι ίδια, ταυτόσιμη. Bene, Καλώς. Και για τη δεύτερη αυτή έκθεση λοιπόν ισχύουν αυτά που είπαμε για την πρώτη. Παραπέμπεται στην αρμόδια Επιτροπή. Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, συνεργασία και περνάμε στην εξήγηση ψήφων. Sulla relazione dell'onorevole Busuttil